Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je vous invite Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Αρχίζει η συνεδρίασή μας της Επιτροπής προεπολογισμών. Σας καλώ να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη πρώτα. Για λόγους τώρα διαθεσιμότητας, θέλω να διευκρινίσω ότι στο σημείο 4 που είναι η εξέλιξη των ε, εργασιών της ομάδας υψηλού επίπεδου όσον αφορά τους ίδιους πόρους, να το εξετάσουμε στις 10 και 30. Γιατί τότε θα είναι διαθέσιμος και κλειμένοι μας ο κ. Λαμασούρ, για παράδειγμα, και ο κύριος Καλφέ. Συμφωνείτε? Καλώς. Τώρα, θέλω να σας ε, μεταφέρω κάποιες πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, μετά από τη σύνταξη του δημοσιονομικού κανονισμού που ολοκληρώθηκε το μήνα που μας πέρασε. Το Κοινοβούλιο έχει πάρει δύο κατεξουδότηση πράξεις που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών και Ελέγχου Προϋπολογισμού τις έχουν ε, λάβει για να αποφανθούν. Τις έχετε κι εσείς. δημοσιεύθηκαν εξάλλου και στο newsletter μας. Και υπάρχει και επιστολή της κυρίας Γεώργεβα η οποία ζητάει από το Κοινοβούλιο να ακολουθήσει μία γρήγορη διαδικασία μη ένστασης της παραγράφου 5 σημείο 6. Για τις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές έχουμε ως προθεσμία την 20 η Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Συνεπώς, θα σας προταθεί μέσω γραπτής διαδικασίας και σε συμφωνία με την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού σύσταση προ αυτή την κατεύθυνση για να υποβληθεί το Δεκέμβριο στην Ολομέλειά μα. Ο στόχο μα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι να αρχίσει 1η Ιανουαρίου του 2016, να αρχίσουν να ισχύουν και έτσι να μπορέσει να εφαρμοστεί πιο εύκολα η μεταρρύθμιση για ολόκληρο το δημοσιονομικό έτος. Είσαστε ενήμεροι λοιπόν για τις κατεξοδότες αυτές πράξεις. Παρατηρήσεις. Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω και για τις αποφάσεις που πήραν οι συντονιστές στις 28 Οκτωβρίου. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την κατανομή των εκθέσεων, αλία, για, με την Μαυριτανία, οι σοσιαλιστές, αληφτική συμφωνία με την Λιμπέρια, το ΕΛΚ. Employee Report για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το δυναμικό τους μια που αυτές συνεισφέρουν ε, σημαντικά στην ανάπτυξη και την απασχόληση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γκουε παίρνει αυτή την έκθεση για τα σχέδια εκθέσεων πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή Ανάπτυξης, η ΝΤΕΒΕ, παίρνει την έκθεση για τις μεταφορές στην Αφρική. Πρόκειται για το άρθρο 55 ή 54, μάλλον το 54 θα ισχύσει τελικά. Έλεγχη τώρα τη σύνθεση ε, τη ομάδα εμπειρογνώμων τη Επιτροπή. Έχουμε γνωμοδότηση από τη δικιά μα την Επιτροπή. Έκθεση έλεγχου προπολογισμού χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων από τον κοινοτικό προπολογισμό. Εδώ θα ζητήσουμε βάσει του άρθρου 54 να είναι κοινή. Ε, προπολογισμοί, δυνατότητε τη Ευρωζώνης και συνέπειε του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού Κοινοβουλευτικός Έλεγχος. Η Επιτροπή μας θέλει συνεργασία με την ΕΚΟΝ βάσει του άρθρου 54. Θα το ξανασυζητήσουμε αυτό αργότερα και με τους συντονιστές. Τώρα, όσον αφορά τις ακροάσεις. Ακρόαση για τα νέα δημοσιονομικά μέσα και τον ρόλο των δημοσίων τραπεζών υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεχόμαστε εδώ συνεργασία με την Ήτρα η οποία την επιθυμεί. Όσον αφορά τώρα αποστολές και αντιπροσωπείες, για την αντιπροσωπεία μας που θα πάει στο Λίβανο και στην Ιορδανία. Εδώ καλούμε τον εισηγητή της ΛΥΜΠΕ να συνοδεύσει την αντιπροσωπεία μας. Αυτές είναι οι πληροφορίες που ήθελα να σας μεταφέρω. Έχετε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 28 και 29 30 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου, 22 Οκτωβρίου. Παρατηρήσεις εγκρίνονται λοιπόν. Και τώρα θέλω να σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα της συνδιαλλαγής όπως γνωρίζετε, πέντε μέρες πριν από την προθεσμία, γιατί έχουμε 21 μέρες μετά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια όσον αφορά το σχέδιο προπολογισμού. Καταφέραμε λοιπόν σε αυτό το διάστημα ε, την Παρασκευή 13 του μηνός να κλείσουμε. Πιο συγκεκριμένα θα έλεγα ότι ήταν το Σάββατο, γιατί ήταν μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Ο Υπουργό Γκραμένια Οικονομικών του Λουξεμβούργου, που προείδρευε τη αντιπροσωπείες του Συμβουλίου, είχε εκδηλώσει την επιθυμία η Παρασκευή αυτή να ήταν μια χαρούμενη Παρασκευή, αλλά βέβαια δυστυχώ εξαιτία των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στο Παρίσι, θα μείνει σαν μια μαύρη Παρασκευή στο μυαλό μας και για τη Γαλλία και για την Ευρώπη ολόκληρη. Και ως ε, εκλεγμένος στη Γαλλία Ευρωβουλευτής, θέλω να σας πω ότι ε, πραγματικά μείναμε όλοι παγωμένοι. Όλοι οι συνάδελφοι που συμμετείχαμε στην συνδιαλλαγή την Παρασκευή το βράδυ και θέλουμε εμεί οι Γάλλοι να σα ευχαριστήσουμε για την αλληλεγγύη σα. Είναι αλήθεια ότι οι τρομοκράτε ε, επιτιθέμενοι με τέτοια δειλία και με τόσο βάρβαρε πράξει επιτέθηκαν στη Γαλλία αλλά και στην Ευρώπη ολόκληρη και στις αξίες μας, στον τρόπο ζωής που έχουμε υιοθετήσει στην Ευρώπη. Ένιωσα λοιπόν αυτή την αλληλεγγύη των συναδέρφων εκείνες τις στιγμές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στη συνδιαλλαγή αυτή και να χαιρετήσω τον Ζαν Μανουέλ. Ήταν μια dream team Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον γενικό μας εισηγητή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ζεράρ Ντεπρέ, ο οποίος παρουσίασε και υποστήριξε τον προπολογισμό για τα άλλα τμήματα. Τον ε, Γιάννη Σκεγέρ επίσης, ο οποίος ήταν... Είναι μόνιμος εισηγητής για τους οργανισμούς και θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τον Τίνεντερ που παρουσίασε τον διαφορετικό προπολογισμό 8 για το 2015 και που έχει άμεση σχέση με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι χώρες μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2016 εξαιτίας του προσφυγικού και της υποδοχής των προσφύγων. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη λοιπόν της αντιπροσωπείας. Είμαστε ανελέγγυοι μεταξύ μας και μπορώ να πω ότι πετύχαμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ακόμα και αν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε χτες σε μια συνάντηση που έγινε στις Βρυξέλλες ότι ο ευρωπαϊκός παραπολογισμός είναι μέτριος και ότι είπε πρέπει να παγιωθεί ο προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών για να σταθούμε στο ύψος των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να προχωρήσουμε καλύπτοντας υποχρεώσεις και τις προκλήσεις. Το πολιετές πλαίσιο είχε καταστεί άκαμπτο. Δεν μας δίνει τα περιθώρια ευελιξίας που επιθυμούμε στην περίπτωση που έχουμε μια μεγάλη κρίση όπως αυτή του προσφυγικού. Συνεπώς, η ενδιάμεση αναθεώρηση θα αποτελέσει μια πολύ σημαντική στιγμή για την Επιτροπή μας και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολόκληρο η Ευρώπη θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις θεμητές προσδοκίες των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ επίσης όλους τους συνεργάτες της Επιτροπής Προπολογισμών. Ευχαριστώ τους πολιτικούς συμβούλους των ομάδων. Ευχαριστώ το σύνολο των υπηρεσιών που μας βοήθησαν σε αυτό το έργο και θέλω εδώ να αναφέρω ιδιαίτερα στους μεταφραστές και τις μεταφράστριες, λέει ο Πρόεδρος. Κάναμε όλοι μαζί μια πάρα πολύ καλή δουλειά και το αποτέλεσμα το οποίο πετύχαμε, αναμφίβολα, είναι το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμούσαμε, που προσδοκούσαμε ένα δις 500.000 επιπλέον και για υποχρώσεις και για πληρωμές σε σχέση με αυτό το οποίο στην πρώτη του εκδοχή είχε αποφασίσει το Συμβούλιο. Αυτό όμως που επίσης πετύχαμε, γιατί η Λουξεμβουριανή Προεδρία ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική, πως ηγήθηκε δηλαδή των συζητήσεων ε, της διατησίας χωρίς φοβερές καθυστερήσεις. Ε, λοιπόν, το αποτέλεσμα μπορώ να σας πω ότι είναι στο ύψος των ελπίδων μας, των προσδοκιών μας. Την επόμενη εβδομάδα θα πάμε στην Ολομέλεια και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τον προπολογισμό αυτό. Είναι μια συμφωνία Έχει να κάνει 555 δισεκατομμύρια στις υποχρεώσει και 144 δισεκατομμύρια στις πληρωμέ. Η Επιτροπή μας δεν ε, χρειάστηκε να αποφανθεί για τα αποτελέσματα της διαλογής αυτά καθε αυτά. Πρόκειται για την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συνδιαλλαγή. 24 Νοεμβρίου θα ζητηθεί και 25 Νοεμβρίου θα έχουμε την ψηφοφορία. Η η Επιτροπή μας θα ψηφίσει για τρία κείμενα μετά από την συμφωνία στη συνδιαλογή. Το διορθωτικό αριθμός 8, το μέσο ευελιξίας και την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Ο Γενικός Συζητητής τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για όσα πετύχαμε την Παρασκευή της 13 του μηνός. Ήταν η μέρα των ε, επιθέσεων των δηλών αυτών στο Παρίσι. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να εργαστούμε σε πνεύμα αλληλεγγύης. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι αυτό που συνέβη στο Παρίσι ήταν μια επίθεση κατά των αξιών όλων μας. Όλοι θα μπορούσαμε να ήμασταν εκεί στο Παρίσι εκείνο το βράδυ. Και η επίθεση αυτή μπορεί να εκλειφθεί ως προσωπική επίθεση από όλους μας. Όλοι θα πρέπει να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς τον γαλλικό λαό. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα θα πρέπει να είναι ε, θα πρέπει να δρά και όχι να περιμένει και να αντιδρά. και πρέπει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για αυτές τις φρικαλαιότητες που διεπράχθησαν στο Παρίσι. Δεν θα πρέπει να ακολουθούμε τα γεγονότα, θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Τώρα, Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τη συνεισφορά τους, χάρη στην οποία καταλήξαμε σε θετικά αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ήταν επιτυχής η προσπάθεια αυτή, παραμείναμε ενωμένοι, είχαμε σαφή στρατηγική. Αυτό που πετύχαμε ήταν θετικό, διότι όλοι όσοι μίλησαν στην αντιπροσωπεία εξέφρασαν μια θέση, η θέση μας ήταν ενιαία, έχουμε έναν προϋπολογισμό για την απασχόληση, για τις εταιρείες και κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουμε και προπολογισμό και κονδύλια και για την επιχειρηματικότητα. Αν δείτε το κεφάλαιο 1α, εκεί αντιστρέψαμε τη θέση του Συμβουλίου στην κατηγορία αυτή και αν δείτε για το 2020 καταφέραμε να ε, αντιστρέψουμε κάποιες από τις περικοπές που επιθυμούσε το Συμβούλιο και έτσι μπορούμε να δώσουμε κάποιες οικονομικές εγγυήσεις που θα στηρίξουν το σχέδιο Juncker. Και έχουμε, όπως σας είπα, και κονδύλι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καλύτερο ε, προπολογισμό για το πρόγραμμα Εράσμους, έχουμε περισσότερα χρήματα για το κόσμο, έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε να διαθέτουμε χρήματα περισσότερα για το Εράσμους, έχουμε και άλλα κονδύλια για την αλληλεγγύη, εσωτερική αλληλεγγύη και εξωτερική αλληλεγγύη. Για μία ακόμη φορά θέλω να πω ότι έχουμε κονδύλια για την αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κονδύλια για θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταφέραμε να περιορίσουμε τις προτινόμενες περικοπές και μη λησμονείτε ότι 97% των τροπολογιών μας αφορούσαν τους δύο βασικούς μας στόχους Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη λοιπόν της αντιπροσωπείας και όλους ιδιαίτερος να ευχαριστήσω τον Ζεράρ Ντεπρέ ο οποίος έκανε πραγματικά έξοχη δουλειά σαν μέρος της ομάδας ένας από τους συνεισηγητές που υπευθύνους ε, για τον προπολογισμό και για το γενικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ήταν δυσχερέστατο το έργο του και τα κατάφερε εξαιρετικά. Επίσης, έχουμε εξαιρετικό εισηγητή για τις υπηρεσίες, τον κύριο Γκάιερ, χάρη σε αυτόν. Προχωρήσαμε, ευχαριστώ και τα μέλη του προσωπικού που μας υποστήριξαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον προπολογισμό του 2015 και το διευθυντικό προπολογισμό υπαριθμών 8. Ήταν η κατηγορία 1α. Για την κατηγορία 1β υπήρξαμε επιτυχής για την κατηγορία 2 πετύχαμε να έχουν περισσότερα για τους γεωργούς και όσον αφορά την κατηγορία 3 κινητοποίησαμε το εργαλείο ευελιξίας το περιθώριο της ευελιξίας στο μέγιστο 1,5 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω και το ίδιο για την κατηγορία 4 που έχουμε 24 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω άρα για τις κατηγορίες όπου είχαμε προτεραιότητες συγκεκριμένες καταφέραμε να χρησιμοποιήσουμε το περιθώριο ευελιξίας επιτυχέστατα. Αυτό ήταν επικοδομητικό για την πρωτοβουλία, για την νεολαία και την απασχόληση και να μην λησμονούμε ότι τα τρία θεσμικά όργανα θεωρούν την απασχόληση των νέων ως ε, προτεραιότητα. Και σε αυτό τον προπολογισμό είμαστε ανοιχτοί για περισσότερες προτάσεις που θα μπορούσαν να υποβληθούν μετά από την αναθεώρηση της ε, πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Τώρα είναι δυνατόν να υποβληθούν και νέες προτάσεις υπό το φως των συμπερασμάτων που, ε, στα οποία καταλήξαμε μετά από την αξιολόγηση για την πρωτοβουλία για την απασχόληση της ε, νεολαίας. Όπως σας έλεγα λοιπόν, στον προπολογισμό αυτό έχουμε σειρά σαφών πρακτικών μέτρων. Ένα είναι που μας απασχολεί, είναι η απασχόληση των νέων, λαμβάνουμε σχετικά μέτρα για την ενίσχυση της απασχόλησής τους και υπάρχει και ένα άλλο πολιτικό μήνυμα που βγαίνει από την όλη προσέγγιση ότι η αναλήψη υποχρεώσεων ε, είναι εκεί για να χρησιμοποιηθούν. Έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις που θα διατηρήσουμε που εμπεριέχονται στο ε, πρόγραμμα Juncker. Γνωρίζουμε βέβαια ότι έχουμε και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για το εγγύς μέλλον και τον ορίζοντα 2020 ε, και το μέσο για τη διασύνδεση της Ευρώπης. Πιστεύουμε ότι αυτά τα προγράμματα τα οποία χρησιμεύουν σαν βάση για το Ευρωπαϊκό Στατικικό Επενδυτικό Ταμείο, μάλλον το, ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων, δείχνει ότι έχουμε πρόβλεψη σωστή για την περίοδο 2014-2020 όσον αφορά τα απαιτούμενα κονδύλια. Όσον αφορά το μέσο για τη διασύνδεση της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι δεν χρειαζόμαστε περισσότερα αρχικά ποσά από τώρα μέχρι το 2016. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε κυρίως όσον σε σχέση με την αναθεώρηση του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου, την ενδιάμεση αναθεώρηση διότι υπάρχουν προγράμματα προς ενίσχυση σε αυτό το τμήμα. Σε όλη τη διαδικασία καταρτήσεως του προπολογισμού κατέστη σαφές ότι στηρίζουμε τη διοργανική συμφωνία, με άλλα λόγια μπορούμε να αυξήσουμε κατά 10% κατά 10% να το αυξήσουμε κατά 10% να το μειώσουμε κατά 10% συμφέρον μας όμως είναι να αυξηθεί ο προπολογισμό για προγράμματα που θεωρούμε σημαντικά. Όσον αφορά τα ποσά που περικόπτονται από το Συμβούλιο και για τις πληρωμές, έχουμε τα πιλωτικά προγράμματα, τα έχουμε ακόμα. Αν δείτε την κατηγορία 5, που θα την παρουσιάσει ο Ζεράρ Ντεπχέ, και το θέμα των υπηρεσιών των ευρωπαϊκών. Τώρα, αν κοιτάξουμε τις πληρωμές, απορρίψαμε τις προτινόμενες περικοπές του Συμβουλίου σε μεγάλο ποσοστό μας υποστήριξε αυτή την προσπάθεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, πιστεύουμε ότι έχουμε σειρά κονδυλίων του προπολογισμού που είναι επαρκή, αλλά θα πρέπει να επαγρυπνούμε. Το 2016 τι θα γίνει με το θέμα των πληρωμών. Θα πρέπει να προσέχουμε τι γίνεται, τα τεκτενόμενα και θα πρέπει να παρενοχλούμε συνεχώς επ' αυτού την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί για μία ακόμη φορά ε, ε, ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι υποχρεώσεις, οι υποχρεώσεων θα πρέπει να υλοποιηθούν και έτσι θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ τους δύο εισηγητές, ευχαριστώ όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας, ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής, όλων των πολιτικών ομάδων, ευχαριστώ τη Γραμματεία, για την έξοχη δουλειά που έκανε κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας και όλος ιδιαίτερος ευχαριστώ τον Αρή Γκυγιόμ ο οποίος μας υποστήριξε σε όλη τη διαδικασία. Πολλά ευχαριστώ στην ε, γραμματεία διότι το προσωπικό είναι υψής της ποιότητας το προσωπικό της γραμματείας διευκόλυνε αφάνταστα τη δική μου δουλειά και του συγητού. Ευχαριστώ το προσωπικό των πολιτικών ομάδων, τους πολιτικούς συμβούλους, όλους και ευχαριστώ ιδιαίτερος τους πολιτικούς συμβούλους του ΕΛΚ, Φάνη, Άννα, Νικόλ, που εργάστηκαν εκατοντάδες ώρες για μας. Φτάσαμε στο τέλος μια, ενός σταδίου των προσπαθειών μας, των εργασιών μας και για μια ακόμη φορά σας λέω ένα ευχαριστώ. Merci, monsieur le Ευχαριστώ κύριε Γενική Εισηγητά. Ε, κύριε Ντεπρέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα, μετά από τις ευχαριστίες του Γενικού Εισηγητού κύριο Φερνάντες και τους επένους που με επιδαψίδευσε, δεν θα ήθελα να μιλήσω και πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος όσον αφορά τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Γνωρίζετε ότι είχαμε ένα στόχο να διατηρήσουμε δηλαδή εκτός της περιμέτρου στην οποία εφαρμόζεται η μείωση το δυναμικό των πολιτικών ομάδων. Το επιτύχαμε αυτό έστω και αν οι άλλες ε, ε, άλλοι, τα θεσμικά όργανα δηλαδή δεν δέχτηκαν να κωδικοποιήσουν ε, την διατύπωση αυτή σε κείμενο σε ό,τι αφορά τις πρόσθετες θέσεις που είχαν ζητηθεί για την ασφάλεια, για τον έλεγχο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έχουμε και την διαχείριση των αποζημιώσεων ε, γραμματείας, όπως λέγονται, ε, είχαμε ζητήσει 48 θέσεις, λαμβάνουμε 39. Το ίδιο για τις προθεσμίες. Για την μείωση τώρα του 5% έχουμε Ουδετεροποιήσει το 2013, αρχίζουμε λοιπόν το 2014, η δε επαλήθευση για το 100% θα φτάσει το 2019. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ε, σωστό το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε. Θα ήθελα τώρα, εξάλλου, για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να μην έχουν γίνει η, 20, η μείωση 20 οργανικών θέσεων. Η απόφαση αυτή δεν είναι σόφρον και στο μέλλον θα χρειαστεί να διορθωθεί. Λίγα λόγια τώρα για την μείωση 5%. Εξετάζοντας τους προϋπολογισμούς των άλλων θεσμικών οργάνων και τα οργανογράμματά τους, διαρωτώ με αν είναι σωστά Αυτές αυτές οι σημειώσεις. Κοίταξα τα νούμερα και νομίζω ότι είναι αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Γεωργίευα. Κάνει προσπάθεια μείωσης μείωση του, του δυναμικού. Έχουν όμως 6.041 συμβασιούχους υπαλλήλους που ισοδυναμούν σχεδόν με όλο το προσωπικό του κοινοβουλίου. Αυτό λοιπόν ε, το 5% αναφέρεται στους ε, μονίμους υπαλλήλους και πάνε να διορθώσουν με τέτοια, να δηλαδή, με, με τέτοια μέτρα. Βρίσκω ότι πραγματικά αυτό δεν είναι αποδεκτό. Για το 2,4% γνωρίζετε ότι εκεί ευνηδιαστήκαμε. Αντί δηλαδή της εφαρμογής ποσοστού προσαρμογής στον τιμάριθμο των μισθών που είχε αρχικά προβλεφθεί. Δεχθήκαμε τελικά ένα 2,4 γιατί βεβαίως η μέθοδος ε, υπολογισμού περιλαμβάνει μάλλον περιλαμβάνεται στο καταστατικό νομίζω στα 64-65 ενώ για του χρόνου κάθε ένα από τα θεσμικά όργανα θα χρειαστεί να κάνει μια προσπάθεια πρόσθετη για να αντισταθμίσει την αύξηση αυτή η οποία δεν έχει εγγραφεί στους προϋπολογισμούς που ψηφίσαμε. Ευχαριστώ και εγώ κατά τα άλλα. όπως ε, και εσείς και ο κύριος ε, Φερνάντες. Ευχαρίστω ο κύριος Φερνάντες τους πάντες, εκτός από τις και τους διερμηνείς. Το κάνω εγώ λοιπόν. Τέλος για τα τραγικά γεγονότα του Παρισιού που δυστυχώς συνέβησαν τη νύχτα εκείνη των διαπραγματεύσεων. Θυμούμε εκείνες τις ε, τρομερές στιγμές όταν αρχίσαμε δηλαδή να συνειδητοποιούμε ε, ποια ήταν η πραγματικότητα που συνέβαινε στο Παρίσι. Βεβαίως σας εκφράζω ε, την συμπάθειά μας και βεβαίως θα μπορούσε να έχει συμβεί σε οποιαδήποτε χώρα. Και σε όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα το Βέλγιο δεν στερείται ευθυνών. Δηλαδή το κατανοούμε αυτό και όλη η ε, πολιτική τάξη του Βελγίου ότι είναι ανάγκη να ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα και σας διαβεβαιώ ότι θα το πράξουμε. Σας ευχαριστώ λέει, ο Πρόεδρος για τα λόγια σας αυτά και η Γαλλία πέρασε τις δραματικές αυτές τις στιγμές βεβαίως τη, τη νύχτα της Παρασκευής αλλά θυμούμε και άλλες χώρες όπως η Ισπανία, όπως το Λονδίνο και άλλες βεβαίως. Ας συμπαραταχθούμε λοιπόν απέναντι στην τρομοκρατία και ας μην υποχωρήσουμε για να την αντιμετωπίσουμε, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές. Κύριε Γκάιερ, εσείς τώρα για τους οργανισμούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα λοιπόν λίγα σχόλια για την διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Ο κύριος Φερνάντες ήδη έκανε την επισκόπηση, έκανε την σύνοψη αυτή που τη βρήκα αρκετή, αρκετά πλήρη. Δεν έχω λοιπόν να προσθέσω τίποτε, ούτε και στις ευχαριστίες που εξέφρασε. Ωστόσο είναι θετική η διαπραγματευτική ε, πορεία μας έως τώρα. Το, η διαπραγματευτική ομάδα αποδείχθηκε άξια και πολύ άξιος εισηγητής ο κ. Φερνάντες. Διότι σε όλη τη διάρκεια της ε, ασκήσεως ε, των καθηκόντων του υπήρξε εισηγητής ολόκληρου του Κοινοβουλίου. Το τονίζω αυτό, δεν ήταν μόνο της πολιτικής του ομάδας. Έτσι κέρδισε την εμπιστοσύνη όλων των συναδέλφων του και με μεγάλη χαρά σας υποστηρίξαμε. Ως σκιώδης ηγητής των σοσιαλιστών σας ευχαριστώ ιδιαίτερος και ελπίζω, εάν αναλάβει η ομάδα μου την εισήγηση για το προπολογισμό του 2017, ελπίζω να μπορέσω να φτάσω και εγώ τον πύχη, αν αναλάβω εγώ δηλαδή για λόγω της ομάδας μου, να φτάσω και εγώ τον πύχη που τον βάλετε υψηλά. Ευχαριστώ και τον κύριο Ντεπρέ. Τα όσα επιτύχατε υπέρ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματικά έφτασε στα άκρα των όσων θα μπορούσε να επιτύχει κανεί. Το κάνατε με ε, εξαιρετική ικανότητα. Έχουμε και εδώ την δύσκολη αυτή κατάσταση όπου το Συμβούλιο για την 5% μείωση του προσωπικού μας επίεσε πάρα πολύ. Νομίζω όμως ότι είχαμε τον σωστό άνθρωπο στη σωστή θέση. Αξίζεται λοιπόν τα συγχαρητήρια όλη τη Επιτροπή Προβολισμού και τα δικά μου βεβαίω προσωπικά. Για του οργανισμού τώρα, η εικόνα εδώ είναι ανάμεικτη. Ω κοινοβούλιο παρακολουθούμε την ε, στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το redeployment pool που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Αυτό προβλέπει ότι ο στόχος της μείωσης κατά 5% του προσωπικού επιβάλλεται ατομικά στον κάθε οργανισμό. και πρέπει να γίνεται αντιστάθμιση αύξησης προσωπικού σε κάποιο οργανισμό με μείωση προσωπικού σε κάποιον άλλο εφόσον τροποποιούνται τα καθήκοντα κάποιου οργανισμού. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα δυσχερές διότι είναι μεγάλος ο αριθμός των οργανισμών που διαθέτουμε, ορισμένοι μάλιστα θεωρούν ότι είναι προβολικά μεγάλος, πάντως έχουν οι οργανισμοί αυτοί αναλάβει ιδιαίτερα καθήκοντα που τους αναθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιος που εργάζεται στον οργανισμό Αλία στο Βίγο δεν μπορεί να πάει ξαφνικά να δουλέψει στον οργανισμό για την ισότητα των φύλων. Είναι λοιπόν εξειδικευμένα πρόσωπα αυτά και σε εξειδικευμένες θέσεις. Πρόκειται άλλωστε για οργανισμούς που είναι αυτόνομοι που αναλαμβάνουν και έξτρα καθήκοντα. Πολλοί ρωτούν πόσους οργανισμούς μπορούμε να καταργήσουμε για να εξοικονομήσουμε χρήματα. Άλλοι όμως έρχονται και λένε να ιδρύσουμε και νέους. Δεν είναι λοιπόν αυτονόητα τα πράγματα αυτά. με αυτό το redeployment pool έχουν φτάσει μειώσεις καμιά φορά σε ορισμένους οργανισμούς και στο 10% και θα χρειαστεί να μειωθούν και άλλοι, να, το προσωπικό και άλλων οργανισμών. Πώς μπορεί όμως να αντιμετωπίσει ένας οργανισμός μείωση κατά 10% του προσωπικού του εάν δεν αυξήσει από την άλλη μεριά την παραγωγικότητα των υπολείπων. Αυτό όμως δεν είναι αυτονόητο, δεν είναι μηχανήματα. Πρόκειται συχνά για οργανισμούς που βασίζονται στην τεχνογνωσία του προσωπικού τους. Αυτό το redeployment pool, εν πάση περιπτώσει, κανονικά πρέπει να είναι ιστορία. Διότι με τις 124 οργανικές θέσεις των frontline agencies αυτής, των οργανισμών δηλαδή που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης του προσφυγικού δεν μπορούν να μπουν σε αυτό το redeployment pool. Επομένως οι υπόλοιποι οργανισμοί έχουν λησμονήσει θα έλεγα σιωπηρά το σύστημα αυτό σίγουρα πάντως δεν το θεωρούν ως πανάκια. Το Συμβούλιο βέβαια επιμένει στην παρουσίαση αυτού του στόχου του 5% μειώσεως θα χρειαστεί να το δούμε. Εξήντα πρόσθετες θέσεις λάβαμε για τον Frontex, για Ευρωπόλ και Άσο 30, 30 και 30 δηλαδή, για Eurojust και για τον Οργανισμό Θεμελιωτών Δικαιωμάτων 2. Τα επιτύχαμε αυτά μετά από διαπραγματεύσεις. Ένας οργανισμός όπου είναι αδιαμφισβήτητο ότι αναλαμβάνει και άλλα καθήκοντα, η ΕΣΑ δηλαδή, που είναι αρμόδια για τους ρυθμιστές ενέργειας και για την εφαρμογή της Ενεργειακής Ένωσης, θα λάβει πέντε πρόσθετες οργανικές θέσεις. Υπάρχουν και οργανισμοί που εν μέρη χρηματοδοτούνται από τέλη που καταβάλει η βιομηχανία. European Aviation Safety Agency στην Κολονία 6 θέσεις. European Chemicals στο Ελσίνικη 3. Και αυτή για τα ε, φάρμακα στο Λονδίνο, Medicine Agency, άλλες τρει. Δεν τολμώ βέβαια να το παρουσιάσω αυτό ως επιτυχία Υπάρχουν οργανισμοί που ζήτησαν 30 οργανικές θέσεις και τα θεμελιώνουν αυτά και τους δίνουμε τελικά το 10% από αυτό. Ε, τώρα να έρθουμε να το παρουσιάσουμε και ως επιτυχία δεν είναι πολύ απλό. Λάβαμε πρόσθετα χρήματα για την ε, European Banking Agency στο Λονδίνο πάλι μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι η συναρματική ισοτιμία μεταξύ ευρώ και ε, λίρα στερλίνας διαμορφώθηκε έτσι ώστε να χρειάζεται περισσότερα χρήματα ο οργανισμό αυτό για να εκπληρώσει τα καθήκοντά του. Βεβαίω όλα αυτά αποτελούν επιτυχίε. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την διάθεσή τη να διαθέσει με τη σειρά τη ε, νέε οργανικέ θέσει, αλλά και η προθεσμία, η, συγγνώμη, η προθυμία του Συμβουλίου αντιμετωπίζουν κάποιους περιορισμούς. Εγώ επέμεινα ώστε ο Οργανισμός Ελέγχου Αλίας να λάβει μία πρόσθετη οργανική θέση. Ορισμένοι τα θεωρούν αυτά ψίχουλα και ότι το περιθώριο στην κατηγορία 2 θα έδινε δυνατότητα να διατεθούν περισσότερα. Όμως θεώρησα ότι δεν πρέπει να ανοίξουμε και άλλο μέτωπο μαζί με το προσφυγικό κλπ. Δεν μπορούσαμε δηλαδή να επιτύχουμε πολύ περισσότερα. Αυτά λίγο πολύ σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι οργανισμοί. Επιτύχαμε λοιπόν ορισμένα πράγματα, ωστόσο δεν τα θεωρώ επαρκή, α το πω έτσι. Ευχαριστώ. Είναι όμως μία πρόοδος. Πρέπει να ευχαριστήσουμε το μόνο μου εισηγητή μας γι' αυτό. Έντερ, εσύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουν υποθεί όλα. Σαν γενική αξιολόγηση, όμως, πρέπει να πω ότι το κλίμα της διαπραγμάτευσης ήταν ιδιαίτερα θετικό. Η Προεδρία έδειξε ότι όταν υπάρχει ένας υπουργό ο οποίος γνωρίζει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τον προπολογισμό, γίνονται αλλιώ οι διαπραγματεύσεις. Ήταν πραγματικά πολιτικές διαπραγματεύσεις και δεν χρειάστηκε να τσακωθούμε, να διαφωνήσουμε για μια λεξούλα, θα πρέπει να είναι αυτή ή άλλη. Έτσι εξοικονομήσαμε χρόνο. Η ενότητα επίσης της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου ήταν στοιχείο κλειδί για την θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της ακολούθησε μια πολύ σοβαρή θέση όσον αφορά τις πληρωμές και ξεκαθάρισε στο Συμβούλιο ότι αν πήγαινε πιο πέρα από αυτά που είχε βάλει στις πληρωμές η Επιτροπή θα ήταν ευθύνη του Συμβουλίου πλέον. Οπότε, ε, αντίθετα από τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε, αυτές εδώ ήταν διαπραγματεύσεις τις οποίες πρέπει να θυμόμαστε και να παραδειγματιστούμε από αυτές. Ελπίζω και του χρόνου και τις επόμενες χρονιές να έχουμε την ίδια τύχη με την Προεδρία, με τη Διαπραγματευτική Ομάδα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να έχουμε δηλαδή πάντα τέτοιες θετικές διαπραγματεύσεις. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους στο Κοινοβούλιο, στην διαπραγματευτική μας ομάδα και μετά μόλις μπούμε στο 2016 αρχίσουμε να δουλεύουμε για το 2017 που θα είναι δύσκολος προϋπολογισμός δεδομένου του πλαισίου μέσα στο οποίο δουλεύουμε. Ένα τελευταίο σχόλιο τώρα για το πλαίσιο. Οι διαπραγματεύσεις πήγαν καλά βέβαια τη νύχτα, όμως το μόνο που θέλαμε είναι να γυρίσουμε σπίτι μας και να ανοίξουμε τις ειδήσει, να παρακολουθούμε την κατάσταση. Όμως συνεχίσαμε ενώ συνέβαιναν αυτά που συνέβαιναν στο Παρίσι, συνεχίσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί ακριβώς αυτό που θέλουν οι τρομοκράτες είναι να μας αλλάξουν τη ζωή, να μας αλλάξουν τη δουλειά, τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και δουλεύουμε και να μην προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε κάτω από αυτές τις συνθήκες ήταν πολύ καλό το παράδειγμα που δώσαμε, ότι συνεχίσαμε να δουλεύουμε και πετύχαμε και το καλό αποτέλεσμα που πετύχαμε. Και στην Ισπανία και στη χώρα των Βάσκων, όπως ξέρετε, έχουμε μεγάλη εμπειρία από τρομοκρατία. Είναι δύσκολο να το καταπιεί κανείς, αλλά πρέπει να αντέξουμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα νικήσουμε την τρομοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να δείξουν αλληλεγγύη και να διαθέτουμε τα μέσα διακυβέρνησης που απαιτούνται για να είμαστε αποτελεσματικοί. Ο κύριος Μανκά όμως έχει ζητήσει το λόγο. Μια σύνταμη ανταλλαγή απόψε να έχουμε γιατί η μερίσια διάταξη περιλαμβάνει πολλά σημεία και πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε επιτύχει πραγματικά ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ήδη τοποθετήθηκαν οι συνάδελφοί μου. Νομίζω ότι ήταν μια κοινή προσπάθεια επιτυχής. Εγώ ευχαριστώ βεβαίως όλα τα πρόσωπα που ευχαριστείτε και εσείς, αλλά ευχαριστώ και ιδίως εσάς κύριε Γενική Εισηγητά, διότι υπό την ε, δική σας ηγεσία, στο πω έτσι, επιτύχαμε πραγματικά σημαντικά αποτελέσματα. Είπατε κύριε Πρόεδρε εσείς ότι ένας προεδρεύων του Συμβουλίου δήλωσε ότι η εξυγένση του προϋπολογισμού πρέπει να προωθηθεί ήδη από τώρα. Εγώ θεωρώ ότι έρχονται εδώ τα μέλη του Συμβουλίου και ψάχνουν να βρουν χρήματα για να αντιμετωπίσουν το προσφυγικό στον Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Προπολογισμό. Σε βάρο των πολιτικών συνοχή. Αυτό είναι κίνδυνο που πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Για τις πληρωμές τώρα θα θυμάστε ότι ήδη τον, ε, την περασμένη άνοιξη είχαμε υιοθετήσει ψήφισμα που ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τέλη Μαρτίου να καταθέσει μελέτη, να εκπονήσει δηλαδή και να υποβάλει μελέτη για τις εκκρεμούσες πληρωμές που ανήρχονταν σε περίπου 2 δισεκατομμύρια. Το έγγραφο αυτό το περιμένω ακόμα, θα είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το, το πρόβλημα, το μέγα αυτό πρόβλημα Τώρα, η πρωτοβουλία για την απασχόληση της νεολαίας. Και τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν ότι θα την προωθήσουν. Όμως αυτό δεν ήταν ε, δεδομένο από την αρχή. Στην αρχή δεν ήθελαν να διαθέσουν ένα ευρώ για την υπόθεση αυτή το 2016. Σήμερα έχουν κάνει τη δουλειά τους οι υπουργοί και θα την υποβάλουν, θα υποβάλουν την ε, σχετική μελέτη στην ε, συνάντησή του του Δεκεμβρίου. Μελέτη που αποδείχνει ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ σημαντική. Τώρα ένα, μια παρατήρηση ακόμα για εδώ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουμε αναλάβει την υποχρέωση τα έτη 2017, 18, 19 να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 170 θέσεις. και ο γενικό Γραμματέας Κλάου Βέλε είπε ότι θα το επιτύχουμε. Όμως πρέπει να συνενούμε στι αποφάσεις μας, γιατί είναι δύσκολο να εξηγήσουμε στου ψηφοφόρου μας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εκπλήττει τι υποχρώσεις του. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για τα αποτελέσματα και ευχαριστώ που με επιτρέψατε να συμμετέχω στη διαπραγματευτική ομάδα. κύριε εκτός μικροφώνου. Και εγώ εκφράζω ικανοποίηση για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, να ευχαριστήσω τον Γενικό Εισαγγελέα, τους κοιόδης ηγητές και εγώ ιδιαίτερα ικανοποιήθηκα βέβαια για τα αποτελέσματα εκδορία 2, διότι ήμουν συγγητής για τη μοδότηση για τον προπολισμό για τη Γεωργία. Έχω κάποια ερωτηματικά όσον αφορά το θέμα των εγγυήσεων για τους νέους. Θα πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις ακόμα για την πολιτική αυτή. Χθες ε, ε, συνάντησα διάφορους νέους από τη Γαλλία με τους υπευθύνους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έπρεπε να τους έρθω σε επαφή μαζί τους και με επαφές με τους ντόπιου μπορούμε να περάσουμε τα μηνύματα. Ο καθένας στη θέση του θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει την πολιτική για την εγγύηση για την νεολαία. Να γίνουν, είναι σημαντικό θέμα για όλη την Ευρώπη. Αυτό που ήθελα να πω κλείνοντας είναι ότι οι επόμενοι, προπολογισμοί θα είναι δύσκολοι δυστυχώ. Σε αυτόν τον προπολογισμό ρυθμίσαν προσωρινά σίγουρα τα θέματα τη μετανάστευση, αλλά βλέποντα τα γεγονότα που συνέβησαν και ακριβώ στι 13 του μηνό, δεν θα μπορούμε επιμακρό να αγνοούμε ποιες, ε, τι θα γίνει με την ευρωπαϊκή άμυνα, με τι ευρωπαϊκέ τα θέματα αυτά. Ε, ο επόμενο προπολογισμό λοιπόν θα πρέπει αυτή τη διάσταση να τη λάβει υπόψη διότι σήμερα είμαστε κάπως αδύναμοι όσον αφορά αυτό το σημείο και πολλές ε, επίσης ευθύνες βαρύνουν τη Γαλλία σήμερα. Ο κύριος Μαραγκάλ είναι ο τελευταίος που θα παρέμβει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να εκδηλώσω τα ίδια συναισθήματα που αισθανθήκαμε όλοι κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής. Ήταν πραγματικά ε, βρισκόμαστε στη συνδιαλλαγή και ζούσαμε ένα επεισόδιο φοβερής φρικτής αντιπαράθεσης στη συνδιαλλαγή. Μας έστειλε όμως και ένα μήνυμα. Έδειχνε ότι πόσο μικρή σημασία έχει αυτά που κάναμε εκεί. Δεν είναι ακόμα η Ευρώπη αυτό που θα έπρεπε να είναι. είναι ο πρώτος προϋπολογισμός της Νέας Επιτροπής, της κυρίας Γιώργεβα. Και αυτό το βλέπουμε, φαίνεται. Αν συγκρίνουμε δηλαδή τη φετινή διαδικασία από την περσινή. Και όχι μόνο στην ικανότητα της Λουξεμβουριανής Προεδρίας, αλλά και γενικότερα και της Επιτροπής. Η συζήτηση δείχνει πόσο περιορισμένοι είμαστε στα στενά πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου που εγκρίθηκε για την περίοδο 2014-2020. Η επιτυχία του κ. Φερνάντες είναι βέβαια μεγάλη γιατί μπορέσαμε να εφαρμόσουμε την κοινή λογική στο περιθώριο που μας επιτρέπει το νέο αυτό δημοσιονομικό πλαίσιο. Επιτρέψαμε να χρησιμοποιηθεί όλο το περιθώριο, να χρησιμοποιήσουμε την ευελιξία όσο γινόταν. Οπότε, από αυτή την άποψη η επιτυχία είναι προφανής, αλλά μας δείχνει και τους περιορισμούς και την απόσταση που μας χωρίζει από την πραγματικότητα που όλοι αναγνωρίζουμε ότι απαιτεί περισσότερους πόρους η ικανότητά μας να επηρεάσουμε τον προϋπολογισμό δεν ξεπερνάει το 1% αυτού του προϋπολογισμού, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πραγματικά όρια της δράσης μας είναι πολύ μικρά. Αλλά πάντως εκφράζω και εγώ μια θετική εκτίμηση όσον αφορά την δημοσιονομική διαδικασία. Η Επιτροπή μας πρέπει να δραστηριοποιηθεί, να μιλήσει κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια. Οι πράσινοι θα ψηφίσουν κατά δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει η συζήτησή μας λοιπόν. Πάντως, μια θετική ψήφος δίνεται αντιλαμβανόμενοι όλοι ότι ο προπολογισμό αυτός είναι το πρώτο μόνο μέρος, όπως είπε και στην αρχική του παρέμβαση ο κύριος Αρτού, δηλαδή η πρώτη μόνο σελίδα της πραγματικής συζήτησης για την μεταρρύθμιση του, δημοσιονομικού, του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου που θα γίνει την Άνοιξη. Έχουν συμβεί πολλά από το 2013-2014. Θα σας αναφέρω μερικά μόνο η συσσόρευση της οικονομικής ε, κρίσης, τα προβλήματα της Ευρωζώνης με την Ελλάδα ως σύμβολο, οι συσσωρευμένες διαφορές μεταξύ χωρών ή μεταξύ περιφερειών. Το ευρωπαϊκό το σχετικό πρόγραμμα ακριβώς αυτό συμβολίζει και παρόλα αυτά πάγωσε. Τρίτον, το προσφυγικό και ό,τι αυτό συμβολίζει. Αντιλαμβανόμαστε ότι κρίναμε έναν προπολογισμό στα ανώτατα του όρια, αλλά παρόλα αυτά δεν αρκεί για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του προσφυγικού. Έπειτα, παγωμένες συγκρούσεις. Την Παρασκευή ήταν, το λέω εγώ, επεισόδιο. Ας ελπίσουμε ότι είναι ένα μεμονωμένο επεισόδιο και δεν θα ακολουθήσουν άλλα. Ασφάλεια λοιπόν, άμυνα, αλλά και ένα κοινωνικό πλαίσιο κατάλληλο να μας προστατεύσει. Και πέμπτο, κλιματικές αλλαγές, αυτό που θα γίνει στο Παρίσι, η διάσκεψη αυτή. Όλα αυτά θα πετούσαν ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και όχι την αναθεώρησή του, μια πραγματική αύξηση, μια πραγματική προσπάθεια για να προχωρήσουμε. Θα το συζητήσουμε σε λίγο για τους ίδιους πόρους. Δεν ξέρω αν ζητάμε πολλά, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή που μας φωνάζει ότι πρέπει να το κάνουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Merci. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για ο κύριος Χριστοφόρου τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καταρχήν να ευχαριστήσω για την τιμή πραγματικά να συμμετάσχω στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής όπου εκεί πραγματικά ζήσαμε μια σημαντική επιτυχία για το Ευρωκοινοβούλιο. Ε, η κορυφαία στιγμή του Ευρωκοινοβουλίου είναι ο προπολογισμό. Και αποδείχτηκε ότι το Ευρωκοινοβούλιο απέδειξε όταν είναι ενωμένο και όταν έχει ισχυρή ομάδα εισηγητών και ιδιαίτερα των κεντρικών εισηγητών ότι μπορεί να καταφέρει αυτά που δεν πιστεύει κανένα. Και αυτή η επιτυχία αντανακλά και σε ολόκληρη την Επιτροπή Προπολογισμών και αν με ρωτάτε εμένα, επειδή στιγματίστηκε από τα τραϊκά γεγονότα, το ότι το Κοινοβούλιο ήταν ενωμένο και έδωσε τη μάχη ήταν και ένα ισχυρό μήνυμα. Ότι μπορεί το Κοινοβούλιο να ενωμένο μακριά από μικροπολιτικές κοπημότητες στα μεγάλα ζητήματα να συμφωνεί. Ήταν μια επιτυχία πέραν από τις πιο αισιόδοξε προβλέψεις και πρέπει να το καταγράψουμε. Άρα με σκληρή δουλειά, με σωστούς και ικανούς εισηγητές, μπορεί το Κοινοβούλιο να πάει και πέραν από τις θεωρητικά οριοθετημένες ε, δυνατότητες του. Πραγματικά για μια ακόμη φορά ευχαριστώ για αυτήν την τιμή και γιατί νιώσαμε περήφανοι για την ε, διαπραγματευτική ομάδα και ιδιαίτερα για τους εισηγητές μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Merci. Alors, José Manuel pour... Euh, ευχαριστώ. Χωσέ Μανουέλ για τα συμπεράσματα τα Ευχαριστώ. Ένα λεπτάκι θέλω για να συναγάγω συμπεράσματα. Θα ευχαριστήσω καταρχάς όλους τους συναδέλφους, όλους σας που συμβάλατε στην προσπάθεια αυτή και πρέπει να σας πω ότι και νομίζω ότι θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους ιδιαίτερως τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία και το Λουξεμβούργιο Υπουργό Οικονομικών για τη δουλειά που έκανε και εκείνος και η ομάδα του. Και αυτή συνέβαλα στην επιτυχία. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κατανόησε απολύτως τις προτεραιότητες μας και μας υποστήριξε. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε και πρέπει μάλλον το υπογραμμίσουμε. Για μία ακόμη φορά θέλω να ευχαριστήσω όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ εσάς κύριε Γενική Συγητά. Πράγματι, τα συμπεράσματα αυτά δημιουργήθηκαν, καταλήξαμε σε αυτά σε μια πολύ σοβαρή ατμόσφαιρα με αισθήματα συγκίνησης που αισθανθήκαμε σε εκείνη τη φάση και είδαμε ότι ε, έπρεπε να κάνουμε προσπάθεια να καταλήξουμε κάποιο θετικά ήταν γιατί πιστεύαμε σε αυτό που κάναμε. Και όταν έχουμε πεπιθήσεις και όταν πιστεύουμε κάτι, συνεννοούμαστε. Και ο καθένας ε, έδειξε ότι ήταν υπεύθυνο και ότι ήταν ρεαλιστής στις συνομιλίες. Πρέπει να ευχαριστήσουμε την Προεδρία, την κυρία Γεωργίευα, πρέπει να ευχαριστήσουμε, που κυρίως ε, κάτσε τη θέση της και στήριξε τη θέση της και θέση μας ε, για τις πληρωμές. Ευχαριστώ τον Hans Γκάιερ. Ένα χρόνο στους δύο έχουμε. Αυτό είναι ο ρυθμός των επιτυχιών. Μια χρονιά στις δύο έχουμε επιτυχίες. Θα ήθελα να σπάσουμε λοιπόν αυτή την αλυσίδα, αυτό το ρυθμό όπου οι επιτυχίες εναλλάσσονται με τις αποτυχίες και με τον Hans Geiger εγώ είμαι σίγουρος ότι θα σπάσουμε αυτό τον κύκλο. Ο προπολογισμό που θα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα ε, θα πρέπει τελικά, ελπίζουμε, να αντιστοιχίσει στην εκτέλεση του προπολογισμού και δεν εκπλήσωμε βλέποντας τις περιστάσεις ε, εάν θα υπάρξουν κατά διάρκεια του σχεδιοθωτικά, ε, διορθωτικοί προπολογισμοί το 2016 και μετά τα χρέη και οι πληρωμές ε, σπρώχνουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο όρος ε, χρεών. Και αν μπορούμε να σκεφτούμε ότι δεν θα άσχημα τα πράγματα το 2016, διότι η καθυστέρηση όσον αναφορά τις υποχρεώσεις επιτρέπει κάπως να ανακουφίσουμε τις ε, πληρωμές, δεν θα εκπλησόμουν αν από το 2017 και πέρα τελικά αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ ευαίσθητες καταστάσεις. Συνεπώς καθένας εδώ πέρα θα πρέπει να προσμετρήσει το εύρος που θα έχει συζήτηση που ξεκίνησε με το Συμβούλιο για την Midterm Revision, την ενδιάμεση αναθεώρηση που θα συζητήσουμε. Θα σταματήσουμε εδώ όσον αφορά το σχέδιο προπολογισμού 2016. Ξέρω ότι υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που θέλουν να διακόψουμε σύντομα και ε, είχαμε να ψηφίσουμε στις 9.50 ε, νο, ίσως θα πρέπει να ψηφίσουμε τώρα και μετά να έρθουμε στην έκθεση ε, για το ΣΥΣ για την 6 και μετά πάμε στον κύριο Γαζαμπάλ στην έκθεση του. Αν έχετε αντιρρήσει, έχετε πρόβλημα. Να πάμε πρώτα στο σημείο 6 και μετά στην έκθεση του κύριου Γαζαμπάλ. Αφού ψηφίσουμε. Λοιπόν, ε, αν έχετε την καλοσύνη να βάλετε τις κάρτες σας ε, μέσα στη συσκευή για την ψηφοφορία. Θα κάνουμε μια δοκιμή καταρχήν όσον αφορά την ψηφοφορία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Δοκιμή τώρα, έτσι. ψήφισαν 25. Λοιπόν, πρώτη ψηφοφορία, Διαστατικός υπολογισμό υπαριθμών 8. 2015. Μήπως μπορούμε να ψηφίσουμε ομαδικά τις έξι τροπολογίες του κ. Άσφορτς. Συμφωνείτε. Υπέρ. Υπέρ. Λοιπόν, θετική ψήφος όσον αφορά το σύνολο των έξι τροπολογιών του κυρίου Άσφορτ. Ποιος θέλει να ψηφίσουμε αυτές τις τροπολογίες. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Το σύνολο τώρα του DAB 8, ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινά. Πέρας. Ψηφίζεται με 22 ψήφους, 2 ε, ψήφοι κατά και 2 προχές. έκρισε εννέα κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μετανάστευσης, τρεις τροπολογίες Ashford. Να τις ψηφίσουμε μαζί, τις τρεις τροπολογίες. Έχετε πρόβλημα. Κανείς δεν έχει αντίρρηση, να τις ψηφίσουμε μαζί. Υπέρ των τριών τροπολογιών. Υπέρ των τριών τροπολογιών. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Στο μέσο ευελιξίας λοιπόν, πάνω σε αυτό, ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει. Πέρας. «23 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά, 2 αποχές» κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για, την, για προκαταβολές. Πώς ψηφίζουμε. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 26 ψήφοι υπέρ, μία κατά, δεν υπάρχει αποχή. Η κυρία Γκαρδιαζιαμπάλ για μία σειρά μεταφορών. Κατηγορία 3. Μια στιγμή να βρω τα χαρτιά μου παρακαλώ. Πρόκειται για τι μεταφορέ 31, 33, 34, 37, 38. Ναι, το βρήκα, Πρόεδρε. Πρόκειται για πέντε μεταφορέ. Η πρώτη, η 31, είναι για να ενισχύσουμε τη γραμμή του προπολογισμού του κόσμου με 8,8 εκατομμύρια ευρώ. Η δεύτερη μεταφορά, αριθμός 33, είναι για να ανταποκριθούμε στην κρίση αναδιόμενων κρίσεων. Ουσιαστικά πρόκειται για την ε, ειρήνη 10 ε, εκατομμύρια. Η 34 έχει να κάνει με τις αλληλευτικές συμφωνίες με την ε, Λιβερία και την Μαυριτανία. Είναι η ιδιαιτερότητα εδώ των αλληλευτικών συμφωνιών, γιατί δεν έχουμε καν τη γνωμοδότηση για τις συμφωνίες αυτές, αλλά πρέπει να μεταφέρουμε ένα τμήμα των χρημάτων πριν να υπογραφεί η συμφωνία αυτή. Και υπάρχει επίσης και η μεταφορά 37. Πρόκειται για 1,3 εκατομμύρια ευρώ που πάει στο ERDF. Δεν ξέρω. Είναι για την βαλτική συνεργασία στην βαλτική. European Territorial Cooperation Baltic Sea. Και το 38 αφορά 1,4 εκατομμύρια για τον μηχανισμό επίλυσης. Αυτές είναι οι μεταφορές που προτείνονται. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Προτείνω λοιπόν να υπερψηφίσουμε. Πρόεδρος, καλώς. Αφού λέτε να υπερψηφίσουμε, καλώς. Ευχαριστούμε για την παρουσία. Να ψηφίσουμε μαζί για όλες τις μεταφορές. Έχετε αντίρρηση για τις πέντε μεταφορές. Ωραία, δεν υπάρχει αντίρρηση. Συνεπώς, με ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίες. 24 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται. Τώρα θα δώσω το λόγο την κυρία Αρντόφσκη που αντικαθιστά τον κύριο Ολμάγερ για τις μεταφορές των άλλων τμήματων για το 2015. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Αντικαθιστώ την κυρία Μόνικα Χολμάγερ η οποία χρειάστηκε να είναι σε άλλη επιτροπή που υπάρχει μια πολύ σημαντική συζήτηση. Θα σχολιάσω λοιπόν για τις μεταφορές αυτές εγώ. Πρόκειται για το Ρίτσι. Σας έχει ήδη ενημερώσει η Μόνικα πολλές φορές για τις μεταφορές αυτές. Δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο εδώ. Πρόκειται για έξι μεταφορές και έχουμε ήδη υποσχεθεί να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Μία μεταφορά είναι στο κεφάλαιο 1 βάση του άρθρου 25 και έχει να κάνει με τον Ευρωπαίο Ομπουτσμαν. Και μια μεταφορά είναι για την Επιτροπή την Οικονομική και Κοινωνική, την ΟΚΕ. Κατά την γνώμη μου δεν υπάρχει εδώ πέρα τίποτα το επίβαχο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι για τις μεταφορές αυτές, κυρίως για την Επιτροπή των Περιφερειών, δράτω με τις ευκαιρίες της παρουσίας του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμών κυρίου συναδέλφου Γκράσλε. Δεν ξέρω αν ξέρετε ποια είναι η κατάσταση που υφίσταται όσον αφορά Επιτροπή Περιφερειών και έναν πρώην υπάλληλο οικονομικό ελεγκτή της Επιτροπής των Περιφερειών, το Ρόμπερτ Μακόι. Δεν θέλω να μακρηγορήσω επ' αυτού. Ίσως μετά αν θέλει κάτι να προσθέσει κάποιος επί της καταστάσεως. Ο Ρόμπερτ Μακόι ήταν financial controller, ασχολείται τον έλεγχο που έχει αρμοδιότητα να ελέγχει την ορθότητα της χρήσης των πόρων εντός της Επιτροπής των Περιφερειών και τα πρώτα έτη στις αρχές του 2000 κατήγγειλε τους ανωτέρους τους για κάποιες πρακτικές κακής διαχείρισης απατών όσον αφορά τις, ε, τους πόρους προτείνοντας ότι θα πρέπει να παρέμβει η Όλαφ δίνοντας το υλικό αυτό. Αυτή ε, η συμπεριφορά οδήγησε σε πολύ βίαιη συμπεριφορά των ανωτέρων του ατόμου αυτού ε, και αυτό οδήγησε τελικά στην απομάκρυση του ανθρώπου αυτού από τη θέση του. Πέρα από τις ψυχικές ζημίες, ψυχολογικές ζημίες που υπέστη για αυτού του είδους ε, την κακομεταχείριση που υπέστη ψανοτέρους, το Ευρωκοινοβούλιο στην απαλλαγή του 2013 και μετά στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού ε, ψήφισε μια συγκεκριμένη θέση που, σύμφωνα με την οποία ζητείται από την Επιτροπή των Περιφερειών να σέβεται τις διάφορες αποφάσεις που το Δικαστήριο των Δημόσιας Υπηρεσιών, το ε, EU Service, ε, Public Service Tribunal, έλαβε αποφάσεις. Η τελευταία απόφαση ήταν το 2014 και διατάσσει την πληρωμή πλευράς της Επιτροπής των Περιφερειών των νομικών δαπανών που υπέστη ο Μακόη, συν μια αποζημίωση που αν δεν κάνω λάθος είναι περίπου 20.000 ευρώ. Μέχρι τώρα η Επιτροπή των Περιφερειών όχι μόνο αρνείται να σεβαστεί τις αποφάσεις αυτές και να εκτελέσει τις αποφάσεις, αλλά δεν παρά την παρέμβαση της, της Όλαφ δεν ακολούθησε επαρκείς εσωτερικές διαδικασίες για την προστασία αυτών των ατόμων που καταγγέλουν ατασταλίες ε, και που κάνουν απλώς τη δουλειά τους. Λοιπόν, ε, ζητώ από όλη την Επιτροπή Προπολογισμού να μην ψηφίσει μεταφορές για την Επιτροπή των Περιφερειών μέχρι ότου κανονίσει σωστά αυτά τα πράγματα και ρυθμίσει τη, τη θέση της όπως πρέπει. Καλώς, ευχαριστώ για αυτή την ανακοίνωση. Δεν είναι όμως ε, στη φύση μας δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε την ημερήσια διάταξη. Θα πρέπει να τοποθετηθούμε επί της αρχής ε, για κάθε μία από αυτές τις μεταφορές, λαμβάνοντας υπόψη σχετική σημασία που έχουν. Ε, ε ίσως δεν χρειάζεται να κάνουν ψηφοφορία αν θεωρηθούν ως ψηφισμένες. Αν έχετε αντιρρήσεις για τη μεταφορά όπως η την Επιτροπή των Περιφερειών θα κάνουμε μια εξαίρεση. εν τη αυτή περιπτώσει. κύριε Φερνάντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά εγώ δεν θέλω να αφήσω να πλανώνται αμφιβολίες επί ζητημάτων που μπορεί να είναι ευαίσθητα όσον αφορά αυτά που υπόθηκαν μόλις τώρα. Και επειδή πιστεύω ότι δεν έχουμε πρόβλημα να αναβάλουμε αυτό το θέμα και εφόσον ο Σιγητή δεν μπορεί να είναι εδώ γιατί παρίσταται σε μια άλλη πολύ σημαντική ε, συνεδρίαση. Προτείνω να ψηφίσουμε τα πάντα με την εξαίρεση του συγκεκριμένου κονδυλίου και στην επόμενη συνεδρίαση μπορούμε να έχουμε όλε τι πληροφορίε όσον αφορά το θέμα αυτό και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα καλό τρόπο να προχωρήσουμε και να επικρατήσει η μέγιστη δυνατή ε, διαφάνεια όπω πάντα αυτός είναι και πρέπει να είναι ο στόχος μας. Ευχαριστώ. Η πρότασή σας είναι έξοχη, κύριε Γενική Εισηγητά. Αν δεν ψηφίσουμε όμως σήμερα, οι μεταφορές θα γίνουν αυτομάτως. Καλύτερο θα ήταν να διεξαχθεί μια ψηφοφορία ε, για να υπάρξει αντίθεση στην μεταφορά. Μου λένε ότι αν δεν διεξαχθεί ψηφοφορία, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τη σχετική που έχουν αυτές οι μεταφορές, Alors, c'est un virement pour info ou pas ci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 διότι δεν είναι αλληλένδετα. Αντίθετα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το θέμα που έθεσε ο κ. Τζανί. αν είναι πάρα πολύ σημαντικό δεν μπορούμε. Το ερώτημα δεν είναι δυνατό να μην απαντήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα μετά να επαληθεύσουμε αν το ερώτημα αυτό συνδέεται διότι πρέπει να είμαστε σοβαροί όταν θέτουμε θέματα επιτάπητος. Και αυτό που ετέθη, το ζήτημα, δεν έχει καμία σχέση με τη μεταφορά, δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να τίθεται το θέμα και να τεθεί άλλη στιγμή. Σε αυτή τη φάση δεν έχω πληροφορίες για να μπορέσω να κρίνω αν υπάρχει σχέση ή όχι. Και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει τώρα να μπούμε σε μια συζήτηση, έχουμε το χρόνο να το κάνουμε Ε, Έπρεπε να το είχαμε κάνει πριν ενδεχομένω αυτή την κουβέντα. Και νομίζω ότι αυτά τα θέματα μπορούν να τεθούν σε άλλε επιτροπέ, κυρίω στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Δεν θέλω να μπούμε τώρα σε συζήτηση επ' αυτού, χωρί να είναι παρόν εισηγητή για αυτό το θέμα. Αν πρέπει να ψηφίσουμε, δεν βλέπω σχέση, θα υπερψηφίσουμε. Αν μπορούμε να αναβάλουμε, κάνουμε την αναβολή. Πρόεδρος, πιστεύω ότι είναι δύσκολο να αναβάλουμε. Δεν είναι τεράστιο το ποσό, είναι θέμα αρχής, το οποίο θα πρέπει να διφωτιστεί. Ο κ. Ζανή έθεσε ένα ερώτημα, έθεσε ένα θέμα. Να το εντάξουμε στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Προπολογισμών. Συμφωνείτε κ. Ζανή. Ο κ. Ζανή λοιπόν συμφωνεί. Συμφωνείτε αγαπητοί συνάδελφοι. Όλες αυτές οι μεταφορές που είναι προς ενημέρωση να θεωρηθούν ως εγκεκριμένε άνευ ψηφοφορίας. Συμφωνούμε. Πάμε λοιπόν στις μεταφοράς, μεταφορές συγγνώμη, πρέπει να ψηφιστούν. Εκεί που έχετε τοποθετηθεί θετικός, συνεπώς θα ψηφίσουμε. η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είναι η πρώτη. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 22 με 3 εναντίον μία αποχή. Επιτροπή των Περιφερειών αυτή μπορεί να αναβληθεί. Alors, oui, monsieur, monsieur Depré. Ο κ. Στεπρέ, αν είναι δυνατόν να αναβληθεί αυτό το σημείο, εγώ θα ήθελα να το αναβάλω, αν γίνεται. Γιατί είναι ευαίσθητο σημείο, θα υπάρξουν και παρόμοιες προτάσεις αργότερα. Να εξηγήσω. Όπως απεφασίστη σύμφωνα τη διαδικασία που προανέφερα ότι θα, θα προσαρμιστούν οι αμοιβέ για το 2016 κατά 2,4% αντί 1,2%. Αυτό ε, οδηγεί σε αύξηση του κόστου ε, για όλο τον προπολογισμό των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των θεσμικών οργάνων για το 2016 και το 2015. Για το 2015 όμω μα αφορά, αφορά μόνο το μισό εξάμεινο, διότι η προσαρμογή ξεκινά από τον Ιούλιο. Για το 2016 είναι πλήρες το έτος. Τι προτείνετε λοιπόν εδώ. Προτείνω να κάνουμε μια συσσόρευση, να τα βάλουμε σε ένα κονδύλι που αφορά τα κτίρια, ούτω ώστε να μπορέσουμε από αυτό το κονδύλι ήδη ε, να ε, κάνουμε περικοπές για τα νίκια και για τα κτίρια για το 2016 από τις πιστώσεις που θα είναι διαθέσιμες για το 2015. Πριν μπούμε στην όλη αυτή επιχείρηση θα πρέπει να συζητήσουμε εδώ διότι ε, νομίζω ότι πρέπει δεν ξέρω κατά πόσο είναι και πιο καλή προσέγγιση που μπορούμε να ακολουθήσουμε πλευρά δημοσιονομικού κανονισμού νομίζω ότι ε, μιλάτε για διακοσμητική ε, άσκηση ε, στα τέλη του Να πληρώσουμε, να κάνουμε τις ώρες, να πληρώσουμε τα νίκια του 2016-2015 και να κάνουμε πιστώσεις για τις αυξήσεις των μισθών χωρίς να φαίνεται. Αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι και ειλικρινείς και να είμαστε υποδειγματικοί εναντί του κοινού ε, όσον αφορά ε, τους ελέγχους των ε, θεσμικών οργάνων με, με, το οποίο ασχολούμεθα. Συμφωνείτε λοιπόν με την αναβολή. αναβολή. Ολοκληρώσαμε λοιπόν για την πολιτική των κτηρίων. Δεν υπάρχει αίτημα μεταφοράς. Επανερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη. Ήτι. Έκθεση Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η κυρία Γκαρδασαμπάλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σύντομα, είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή αυτή προπολογισμών γνωμοδοτεί στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το 2014. Βασίζω την γνωμοδότησή μου σε τρία σημεία. Πρώτον, το σχέδιο Juncker είναι η πρώτη φορά που κάνουμε μια έκθεση στην οποία μπορούμε να μιλήσουμε για το σχέδιο Juncker. Έπειτα, πρέπει να τηρηθεί το στοιχείο της προσθετικότητας. Πρέπει να το φροντίσουμε αυτό. Και έπειτα υπάρχει η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες και Ιδρύματα. Είναι αλήθεια ότι βελτιώθηκε η ενημέρωση από πλευρία της ε, ΕΤΕ για την χρήση των δημοσιονομικών εργαλείων, αλλά πρέπει να έχουμε και μια συνολική εικόνα που λείπει. Κάτι που να μας επιτρέπει να έχουμε την συνολική εικόνα και έτσι να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε. Φυσικά θέλουμε και λεπτομέρειες, και τα δύο θέλουμε δηλαδή, και τη γενική εικόνα και τις λεπτομέρειες. Επίσης, ζητάμε από την ΕΤΕ να χρησιμοποιήσει ό,τι μέσα έχει στη διάθεσή της για να ενισχύσει τη συμμετοχή των άλλων θεσμικών οργάνων και άλλων τραπεζών για να συμμετέχουν στα χρηματοδοτικά αυτά μέσα. Επίσης, τώρα κάτι που έχει να κάνει με την εξωτερική εντολή. Εδώ πέρα γίνεται μία το εξή. Ζητάμε να ελέγχουμε την εκτέλεση της εντολής και να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι τρία δις είχαν προβλεφθεί από την αρχή για την αναθεώρηση τη μεσοπρόθεσμη να μπορούν όντως να εξεταστούν σαν προσθήκη. Θέλω να υπογραμμίσω ότι όλα τα προγράμματα, όλα τα σχέδια τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές και με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς να μην έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΤΕΠ. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Παρατηρήσεις. Παρακαλώ, κύριο Σταρό. Ε, Ο κύριο συγγνώμη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σύντομα, λίγα σχόλια που ε, θέλουμε να επισημάνουμε εμεί οι πράσινοι και αφού βέβαια εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το ξεκίνημα της λειτουργίας του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, αλλά βεβαίως πρέπει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εξασφαλίσει την προσθετικότητα των ε, κονδυλίων. Διότι εμείς ανησυχούμε ότι πολλά από τα project θα έβρισκαν ε, ε, χρήματα για επενδύσεις ούτως ή άλλως και υπό κανονικές συνθήκες και δεν θα χρειαζόντουσαν άλλα. Εμείς θέλουμε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αναλάβει περισσότερους κινδύνους και να ξεφύγει από αυτή την οτροπία ότι πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει το τριπλό α κάθε επένδυση που θα κάνει. Και να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την συμμόρφωση με τα σχετικά κριτήρια. Δεν είναι βέβαια και άχρηστο να υπενθυμίζει κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είναι και τόσο διαφανής, για να μην πω ότι είναι εντελώς αδιαφανής, άρα χρειάζεται να προσέξουμε πολύ περισσότερο στις πρακτικές που ασκεί για το πώς χρησιμοποιούν οι κυρίες και οι κύριοι αυτής της τράπεζας τα χρήματά μας. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την υποχρέωσή μας να ελέγχουμε την εξωτερική εντολή της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων και την ενδεχόμενη ενεργοποίηση πρόσθετων 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και να εξετάσουμε προσεκτικά την πρώτη έκθεση ολοκλήρωσης έργου και για την εντολή για εξωτερικό δανεισμό για την ε, επόμενη περίοδο. Ευχαριστώ κύριε Τάραντ. Μούρεσαν. Ευχαριστώ και από τη δική μου πλευρά. Ευχαριστίες στην κυρία Γκάρδια Θαμπάλ για τη γνωμοδότησή της που απηχεί την άποψη της πολιτικής μας ομάδας επίσης. Μετά από την θέση ισχύ του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ενισχύεται και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων, όπως θα εξηγεί και η κυρία Κάρδια Θαμπάλ. Τρία σχόλια που δεν έρχονται σε αντίφαση με τα όσα διαλαμβάνει η έκθεση, αλλά που μπορούν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν προσθέτως. Πρώτο, ο ρόλος χρηματοδότησης μικρών και μεσών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα να αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην πρόσβασή τους σε κατάλληλη χρηματοδότηση και η ΕΤΕ μπορεί να αποτελέσει τμήμα της λύσης. Μπορεί να τους βοηθήσει πολύ στους ανθρώπους αυτούς. Και νομίζουμε ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ενισχύσει τα χρηματοδοτικά μέσα, ειδικώ για μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Δεύτερο, η εξωτερική εντολή της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων απέναντι και στις ανατολικές και στις νότιες γειτονικές χώρες της Ένωσης που αντιμετωπίζουμε βεβαίω και πολλές κρίσεις και στην Ουκρανία αλλά και προς Νότον αν όμως θέλουμε να σταματήσουμε τα κύματα ε, προσφύγων προς την Ευρώπη, πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης στις χώρες τους. Εκεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να παίξει ρόλο στην βελτίωση των κοινωνικών υποδομών με επενδύσεις στα αστικά κέντρα, στα συστήματα υγείας, στην παιδεία για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στις πατρίδες τους των ανθρώπων αυτών. Εκεί μπορεί, μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τρίτο, εξακολουθούμε, να βλέπουμε σημαντικές γεωγραφικές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών μελών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων. Να εξετάσουμε λοιπόν προσεκτικότερα πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις γεωγραφικές και διατομιακές ανισότητες με την κατάλληλη χορήγηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και η δική μας ομάδα θα υποβάλει σχετικές τροπολογίες που δεν έχω σε αντίφαση με το κατά τα εξαιρετικό περιεχόμενο της εκθέσεως της κυρίας Γουάρια Ζαμπάλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν βλέπω κανένα άλλος να ζητεί το λόγο. Κατάθεση τροπολογιών μέχρι τις 23 ενδεκάτου στις 5 το απόγευμα. Ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών στις 10 Δεκεμβρίου. έλεγχος προπολογισμού 28 Φεβρουαρίου και ολομέλεια στις, ε, το Μάρτιο. Τώρα, το λόγο ας λάβει ο εισηγητής μας Γιάννης Λεβαντόφσκι καθώς και ο Ζεράλ Δεπρέ. Και αυτό για την διαδικασία, για την προστιθέμενη αξία και για το εθνικό εισόδημα. και την αποτίμηση των πόρων. Ποιος θα μιλήσει πρώτος? Ο Γιάννος. Συγχαρητήρια και προς εσάς και προς όλους εκείνους που είναι πίσω από το θαύμα αυτό για τον προπολογισμό του 2016 υπό εξαιρετικές συνθήκες. Γεράρ και εγώ έχουμε μια τεχνική τροπολογία σε τεχνικό κανονισμό για το πώς να κινητοποιηθούν οι ίδιοι πόροι που συμφωνήθηκε το 2014 για να αρχίσει να ισχύει υποτίθεται από το 2016 αλλά για να εφαρμοστεί και αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2014. Η ιδέα της τροπολογίας αυτής στον κανονισμό είναι να γίνει ο κανονισμός ακόμα πιο τεχνικός ώστε σχεδόν αυτόματα να εφαρμόζεται πέραν πολιτικών επιρροών και εμείς υποστηρίζουμε την ιδέα να γίνει αυτοματοποιημένη η εφαρμογή του. Βασισμένη στην εμπειρία του 2014, υποστηρίζουμε κίνητρα να γίνονται οι καταβολές έγκαιρα. Επίσης να κινητοποιείται ένα παραπάνω δωδεκατημόριο ώστε να αντιμετωπιστεί το συσσωρευμένο χρέος του κοινοτικού προπολογισμού. Επίσης να υποστηριχθεί αυτά τα αρνητικά επιτόκια τα οποία δεν επιτρέπεται να επηρεάσουν τον προπολογισμό. Η μόνη πραγματική λοιπόν τροπολογία, το περιεχόμενο ε, της δηλαδή, έχει ότι έχει εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για το θέμα όχι μόνο στο Συμβούλιο αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι τεχνική τροπολογία και ως τέτοια μπορεί να υποστηριχθεί από όλους. Κύριε Ντεπρέσης. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπε με έξοχο τρόπο συνάδελφός μου ο κύριος Λεβαντόφσκι. Να πω απλώς ότι η εμβέλεια αυτών που θα κάνουμε είναι σχετικά περιορισμένη διότι πρόκειται περί κανονισμού του Συμβουλίου μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Ελεκτικό Συνέδριο. Λοιπόν, εξετάσαμε ο Γιάννους και εγώ το κείμενο. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να το στηρίξουμε με την τροπολογία που προτείνουμε. Πολύ καλά, δεν ζητά κανείς το λόγο. Να σας διευκρινίσω κάτι, ότι οι τροπολογίε θα πρέπει να κατατεθούν τα αργότερα 24 Νοεμβρίου στι 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 3 Δεκεμβρίου και στη δεύτερη ολομέλεια του Δεκεμβρίου θα ε, υπάρξει τοποθέτηση επιστροποποίησης του κανονισμού. Ερχόμαστε λοιπόν στην ακρόαση των φίλων μας της ομάδας υψηλού επίπεδου για τους ιδίους πόρους οπότε θα ζητήσουμε από ε, ε, θα ζητήσουμε να συνεδριάσουμε και κλεισμένων των θυρών. Ζητώ λοιπόν στους επισκέπτες και τους εκπροσώπους των άλλων θεσμικών οργάνων εγκαταλείψουν την αίθουσα σας παρακαλώ και θα σταματήσουμε και τη μετα...